och varmt välkomna till eh, det här återupptagna. Καλημέρα σας. Θα συνεχίσουμε σήμερα τη συνεδρίαση της πολιτικής μας ομάδος. Ξεκινάμε αμέσω με το σημείο 11 της ημερησίας διάταξης και επ' αυτού πρόκειται για συζήτηση και συνεννόηση σχετικά με την ε, ε, αποστολή της Επιτροπής στην Βαρσοβία και οι συμμετέχουσες Πρέπει ίσως να σας πω εγώ, δεν ε, μπορούν να μας ενημερώσουν ε, ε, άλλοι, αλλά εκ μέρους της... Με συγχωρείτε, όχι. Εγώ ήμουν εις την αποστολή αυτή, συναντήσαμε την, τις εκπροσώπους από την κοινωνία των πολιτών και ε, τελικά διαπιστώσαμε ότι δεν συμμετείχαν ε, όλες οι μη κυβερνητικέ οργανώσεις τις οποίες ε, είχαμε ε, καλέσει αλλά μπορέσαμε να συζητήσουμε πώς μπορούμε να βοηθήσουμε τα θύματα της βίας κατά των γυναικών, τα θέματα της υγείας και επιπλέον συζητήσαμε την θέση των γυναικών εις την αγορά εργασίας και επιπλέον συναντήσαμε και ε, το Κογκρέσο των Γυναικών που είναι ε, μία ε, οργάνωση με 200 μέλη είναι η πιο μεγάλη οργάνωση στην Πολωνία με εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών και συνεργάζονται επί διαφόρων θεμάτων με σχετικά ε, ε, με αυτή την οργάνωση βλέπετε ένα σωρό ε, ενδιαφέρουσες γυναίκες με πολλά χαρακτηριστικά και νομίζω ότι η συνάντησή μας με αυτή την εκπροσώπηση ήταν πολύ καλή συζητήσαμε για τις ποσοστώσεις. Αυτό ήταν ένα από τα θέματα της συζητήσεώς μας. Επίσης ε, σχετικά με τη νέα νομοθεσία της Πολωνίας, σχετικά με τις ε, ε, εκλογές και την προεκλογική περίοδο όπου προβλέπεται ότι τουλάχιστον 35% των μελών των εκλογικών καταλόγων που προσφέρονται για εκλογές πρέπει να είναι γυναίκες. Ε, συζητήσαμε και με την Πολωνική Προεδρία. Ε, θυμάστε ότι μας έχουν καλέσει να συμμετάσχουμε στο συνέδριο των γυναικών 17 και 18 Σεπτεμβρίου. Ε, συναντηθήκαμε και με την κυρία Ρατζέσκα που είχαμε χθες εδώ στην συνεδρίασή μας και με αυτήν συζητήσαμε για την ε, νέα ε, νομοθεσία ε, για την κατάργηση των διακρίσεων που ψηφίστηκε το 2010 για το γυναικείο εκλογικό σώμα και επίσης για την κοινωνική πολιτική. Επιπλέον λάβαμε πληροφορίες σχετικά με τις προτεραιότητες της Πολωνικής Προεδρίας κατά τη διάρκεια της θητείας τους και συζητήσαμε και διάφορα άλλα θέματα όπως την οδηγία για την άδεια μητρότητος, ε, για την περίθαλψη των παιδιών, για το τι υπηρεσίες προσφέρονται, ε, το σύστημα της ε, υγειονομικής περίθαλψης. Και η υφυπουργό μας πρότεινε να ξανασυναντηθούμε ε, και να ξανασυζητήσουμε ιδίως την ε, οδηγία της ε, άδειας μητρότητος ε, η οποία θα διεκπαιρεωθεί κατά τη διάρκεια της Πολωνικής Προεδρίας δηλαδή να συναντηθώ εγώ με την εισηγήτρια και τον εκπρόσωπο της Πολωνικής Κυβέρνησης κατά τη συνέχεια μας κάλεσαν για γεύμα στο Κοινοβούλιο και ε, στη συνέχεια είχαμε μία συνεδρίαση με τους εκπροσώπους της ε, Πολωνικής ε, Προεδρίας και τέλος συναντηθήκαμε με άτομα που εκπροσωπούν την Ευρωπαϊκή Ένωση στην Πολωνία στο τέλος υπήρξε μία συνέντευξη ε, τύπου. Αυτά ήταν ουσιαστικά τα θέματα. Ε, υπάρχουν όμως ιδίως δύο που θέλω να συζητήσω. Δεν ξέρω αν ε, κάποιο άλλο μέλος της αντιπροσωπείας θέλει να παρέμβει τώρα, αν υπάρχει κάποιος από εσά ε, που ήταν στην ε, αντιπροσωπεία, αν θέλει κάτι να προτείνει, αν έχει ερωτήματα σχετικά με την επίσκεψη αυτή. Διαφορετικά έχουμε συμπληρώσει και καλύψει το άρθρο 11 και προχωράμε στη συνέχεια της ημερησίας διατάξεως. Οπότε, ερχόμαστε στο επόμενο θέμα. Το επόμενο θέμα είναι το 13, η θέση του Κοινοβουλίου σχετικά με το σχέδιο προϋπολογισμού όπως τροποποιήθηκε από το Συμβούλιο και θα εξετάσουμε όλα τα τμήματα. Η συγγήτρια είναι η κυρία Ματέρα, η οποία είναι η συγγήτρια για γνωμοδότηση και θέλω να σας πω ότι η Επιτροπή μας ήδη έχει τοποθετηθεί ε, σχετικά με ε, το προϋπολογισμό στις 25 Μαΐου. Υποβάλαμε τη γνωμοδότησή μας στην Επιτροπή Προϋπολογισμού η οποία την έλαβε υπόψη και την περιέλαβε στο ψήφισμα του Κοινοβουλίου κατά τρόπον ώστε να έχουμε εντολή για να διαπραγματευτούμε τον προϋπολογισμό του 2012. Τώρα βρισκόμαστε στο επόμενο βήμα και πρέπει να ε, βρούμε ε, τροπολογίες ε, σχετικά με τον προϋπολογισμό του επομένου έτους. Όσον αφορά την αντιπροσωπεία μας, ε, το Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων ε, ε, μας απασχολεί όπως και το πρόγραμμα Δάφνη και επειδή ε, έχουμε ε, τώρα λίγο χρόνο θα δώσουμε τον λόγο ή στην εισηγήτρια την κυρία Ματέρα για να μπορέσει να μας, παρα... μας εμεινερώσει που βρισκόμαστε. Ευχαριστώ. Ως εισηγήτρια για την Επιτροπή των Γυναικών για τον Προϋπολογισμό ως προς τον Προϋπολογισμό 2012 θα ήθελα να σας μιλήσω για τα δεδομένα του Συμβουλίου. Όπως είπατε και εσείς, έγιναν πολύ σημαντικές περικοπές σε σχέση με τον προπολογισμό 2011, σε σχέση με τις πολιτικές ε, ισότητας μεταξύ των δύο φύλων. Είναι σημαντικές αυτές οι περικοπές. Ως προς το Ινστιτούτο του Βίλνιους, είτε και μάλλον και η Επιτροπή και το Συμβούλιο ζήτησαν μείωση κατά ένα εκατομμύριο ευρώ και δυστυχώς δεν θα μπορέσει να λειτουργήσει καλό στο Ινστιτούτο Ισότητας των Δύο φίλων στο Βίλνιους μέσα στα πλαίσια και της Πολωνικής Προεδρίας. Και δεν θα μπορέσει να βοηθηθεί και από τα κράτη-μέλη. Ως προς τα θεμελιώδη δικαιώματα και ηθαγένεια του προγράμματος DAFNE, για την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών υπάρχει μία μικρή αύξηση της τάξης των 300.000 ευρώ ως προς τις πληρωμές. Αλλά και η Επιτροπή και το Συμβούλιο προτείνουν μία περικοπή κατά 2,5 εκατομμύρια ως προς αναλήψεις υποχρεώσεων για το 2012. Εγώ νομίζω όμως ότι θα πρέπει να υπάρχουν ίδιες πιστώσεις που ίσχυαν για το 2011 για το πρόγραμμα DAFNE, γιατί τουλάχιστον το 20-25% των γυναικών στην Ευρώπη έχει τουλάχιστον μία φορά υποστεί βία είτε εντός είτε εκτός σπιτιού. Άρα δεν μπορούμε να δεχτούμε αυτή τη δραστική περικοπή επί ενός προγράμματος το οποίο χρησιμοποιείται κατά πολύ από τα κράτη-μέλη. Δηλαδή αυτή τη μείωση την εκλαμβάνω ως μια βία, μια μορφή βίας κατά της Επιτροπής Γυναικών. Τέλος, ως προς το πρόγραμμα Progress, το Συμβούλιο προτείνει μία μείωση ανάληψης υποχρεώσεων και δαπανών 540.000 ευρώ σε σχέση με το 2011. Εγώ όμως είμαι υπέρ της αρχικής πρότασης Κομισιόν που ήταν της τάξης των 2 εκατομμυρίων ευρώ για το πρόγραμμα Progress για την προώθηση δηλαδή της απασχόλησης, της κοινωνικής ένταξης, έτσι ώστε να βγούμε έστω και αργά από αυτή την οικονομική κρίση. Με συγχωρείτε, δύο εκατομμύρια και όχι δις όπως είπα στην αρχή. Δύο, εγώ είπα δύο δις στην αρχή, ενώ εννοούσα δύο εκατομμύρια, 845.000. Δικό μου το λάθος. Επειδή είμαι και μέλος της Επιτροπής Προϋπολογισμών, μπορώ να πω ότι δεχτήκαμε μεγάλες περικοπές, αλλά ήταν αναπόφευκτο εάν λάβουμε υπόψη τις γενικότερες περικοπές για τις ευρωπαϊκές πολιτικές στον τομέα της ΚΑΠ, της ενέργειας και ούτω καθεξής. Και εμείς ως Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας μεταξύ των δύο φύλων θέλαμε να τύχουμε υψηλότερης υποστήριξης. Όμως συμβαδίζουμε με αυτή τη λιτότητα η οποία μας επιβλήθηκε και ισχύει για ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ελπίζουμε στο μέλλον να μπορέσουμε να βγούμε από αυτή την οικονομική κρίση και να συνεχίσουμε να εφαρμόζουμε τα σημαντικά αυτά προγράμματα για την Επιτροπή μας, αλλά και για ολόκληρη την Ευρωπαϊκή, ε, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κυρία Ματέρα. Η κυρία Μπάουερ. Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω το εξή. Πέσε να συζητήσαμε το του προγράμματος δάχνη Θυμάμαι ότι είπαμε για αυξημένη πρικοδότηση του προγράμματος. Και το πρόβλημα ήταν ότι εκεί είχε εγγραφεί κάποιο ποσό, κάποιο κονδύλιο για 7 χρόνια. Δεν θυμάμαι πόσο ήταν. Και αν γίνει αύξηση για μια χρονιά, αυτό σημαίνει ότι θα έχει λιγότερα την επομένη. Αυτό σας ρωτώ. Τι γίνεται, τι ισχύει όσον αφορά αυτό το πλαίσιο προπολογισμού για το Δάφνη. Και τι θα γίνει για την επόμενη διετία. Τι, τι ποσά προβλέπονται, τι κονδύλια πρόκειται να διατεθούν για το Δάφνη. Θεωρώ ότι σαν συνέπεια της ε, υιοθέτησης αυτής της ε, Σύμβαση στο Σύμβουλο τη Ευρώπη. έχουμε έξτρα κάποια καμπάνια, εκστρατεία τη ε, οπότε και θα χρειαστούν περισσότερα χρήματα του χρόνου περισσότερα πόσα όσα τις προηγούμενες χρονιές Πρόεδρος Σας ευχαριστώ κυρία Μπάουερ Νικολά Έχω μόνο μια μικρή παρατήρηση όσον αφορά τον προπολογισμό του Ιδρύματος για την ισότητα. Έχουμε γεννούργιο θεσμικό όργανο και δώσαμε αγώνα γι' αυτό, οπότε η συρρήκνωση του προπολογισμού είναι κακό σημάδι, ε, ούτως ώστε να μπορέσουμε να έχουμε το ίδιο υψηλό επίπεδο αντιμετώπιση του θέματος ισότητας των ε, φίλων. Νομίζω ότι θα πρέπει να υπάρξει κάποια τροπολογία σε σχέση με αυτό, όλες, όλοι να προσθέσουμε αυτή την τροπολογία, ούτως ώστε να μην σταθερό ο προπολογισμό αυτού του θεσμικού οργάνου. Κύριε Νικολάη, σα ευχαριστώ. Τώρα Ναι, συμφωνώ με αυτό που είπε κύριε Νικολάη. Υπάρχει ε, και ε, είχε εξηγηθεί ότι ο προπολογισμό ε, ήταν εντάξει, αλλά και ακριβώ και εγώ μιλώ για αυτό το ίδρυμα του Βίλνιου για την ισότητα. Ε, το είπε η Μπάρμπαρα, δεν ξέρω, δεν, δεν, δεν πρόσεξα γιατί τι έλεγε στην αρχή. Οπότε είχαμε, πάει, είχαμε πει ότι θα υπάρξει κάποια αύξηση, διότι μέχρι σήμερα είπαμε ότι η κυβέρνηση της ε, Λιθουανίας θα αναλάμβανε την εγκατάσταση και στο μέλλον μια που είπαμε ότι ενδεχομένω αυτό μπορεί να πάει σε κάποιο πιο προβλημένο μέρος, πιο κατάλληλο και έχουμε επίση και την αντιπροσωπεία εκεί και είπαμε ότι πρέπει να γίνει αυξημένη προϋποδότηση γιατί βέβαια τώρα που έγινε αυτή η αλλαγή ε, ε, χρειάζονται περισσότερα χρήματα. Επομένως θα πρέπει να αντιταχθούμε στη σύγκρουση του προπολογισμού και ε, ακριβώς όχι μόνο δεν φτάνουν τα χρήματα σήμερα αλλά ε, ε, θα χρειαστούν περισσότερα. Μια που ακριβώς τώρα πρέπει να πληρωθεί κάποιο μίστομα το οποίο δεν πληρώνονταν πριν. Ευχαριστώ κύριε Ταραμπέλα. Η επόμενη. Γιωμάνη. Συμφωνώ με όλους εσάς ότι η χρηματοοικονομική κρίση έχει κοστίσει γιατί έχουμε τα μέτρα λιτότητας των κρατών μελών και όλο το, όλο αυτό το, σοκ. Αλλά θα σας πω ότι άρχισε η λειτουργία του ιδρυματος δυο δύο-δυόμιση χρόνια αργότερα από τότε που προβλεπόταν. Και παρ' όλα αυτά υπήρχε προπολογισμό που χρησιμοποιείται για άλλους σκοπούς αυτά τα δύο χρόνια. Άρα είναι πάρα πολύ σημαντικό να παραμείνει ο ελάχιστος προπολογισμό που ίσχυε. Είναι πάρα πολύ σημαντικό το θέμα της ισότητας. Δεν είναι δυνατόν να τιμωρούμε την υπόθεση της ισότητας λόγω των μέτρων λιτότητας. Να μην το δεχτούμε, Μπάρμπαρα, δεν ξέρω. Θα μπορούσαμε να αντεβάσουμε κάποιο είδους ε, ε, τροπολογία στην Ολομέλεια. Είναι απαράδεκτη η μείωση. Ένα εκατομμύριο είναι τεράστιο ποσό. Και λαμβάνω. κατά την προετοιμασία, νομίζω το 2009 που ξεκίνησε, δεν ξοδέψαμε δεκάρα. Αλλά δεν ξέρω που πήγαν αυτά τα χρήματα. Εγώ δεν είμαι τόσο σίγουροι ότι πήγε για θέματα ισότητα. Μάλλον είμαι βέβαιο. Άρα για να σκεφτούμε τι θα κάνουμε, γιατί πιστεύω ακράδαντα, ότι πρέπει να προωθήσουμε αυτό το κοινό μας όριγμα που το έχει αριστερά και δεξιά ε, και να μείνουμε σταθεροί στα πιστεύω μας. Σας ευχαριστώ, λέει η Πρόεδρος. Κύριε Φιγκερέδο, ευχαριστώ, Πρόεδρε, και εγώ θα ήθελα να αρχίσω το Ινστιτούτο για την Ισότητα, γιατί φαίνεται ότι πρόκειται για μια μεγάλη περικοπή εδώ. Αν λάβουμε υπόψη και τις δυσκολίες που αντιμετώπισε για να αρχίσει να λειτουργεί και πέρασαν πολλοί μήνες, σχεδόν δύο χρόνια, μέχρι ότου λειτουργήσει ευπρεπώς. Μετά είχαμε δυσκολίες για να λειτουργήσει πλήρως. Και αυτή τη στιγμή με αυτές τις περικοπές δεν μπορεί να ανταποκριθεί στους στόχους, τους, στους στόχους του. Δεν το κατανοώ. Νομίζω ότι η Επιτροπή μας θα έπρεπε να διατρανώσει τη θέλησή της σε σχέση με αυτό το θέμα να ρωτήσουμε την Επιτροπή τι συμβαίνει, υπεύθυνε και το Συμβούλιο για αυτή τη δραστική περικοπή. Και βεβαίως δεν μιλώ μόνο για τις πιστώσεις, αλλά θα πρέπει να είμαστε απόλυτα σαφείς. Επί δεν ξέρω, μπορούμε να υποβάλουμε μια προφορική ερώτηση έφνης. Νομίζω όμως ότι θα πρέπει να ε, αντισταθούμε, να παραπονεθούμε έντονα. Όσον αφορά τις άλλες στήλε, νομίζω ότι ο κοινωνικός τομέας και ο τομέας ισότητας επειδή έχει ε, υποστεί δραστικές περικοπές, πλήττει ιδιαίτερα τις γυναίκες. Δεν χρειάζεται να επιμείνω σε αυτό. Εδώ οι πιστώσεις είναι πολύ ναι, ναι, περιορισμένες ναι, όσον αφορά τις πληρωμές ε, και ως προς το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ή στον τομέα της ισότητας. Δεν είναι... Δεν μπορούμε να παραδεχτούμε, να δεχτούμε κάτι τέτοιο. Δηλαδή ήδη θα έπρεπε να προτείνουμε αυξήσει διότι για ορισμένες χώρες θα έπρεπε να μιλήσουμε για συγχρηματοδότηση, για μεγαλύτερη συγχρηματοδότηση στο κοινωνικό τομέα. Αλλά αυτό δεν μπορούμε να το απαιτήσουμε από οργανισμούς που δεν μπορούν να συμμετάσχουν κατά 20-30% στη χρηματοδότηση. Δηλαδή θα έπρεπε να μειωθεί αυτή η συγχρηματοδότηση. Και αυτό που έχει σημασία είναι να μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε αυτά τα χρήματα κατά καλύτερο τρόπο. Δεν κατανοώ επίσης τι συμβαίνει με το πρόγραμμα Progress ομολογουμένως και θα ήθελα να μου πείτε, να μου δώσετε ορισμένες επεξηγήσεις. Δεν ξέρω κατά πόσο έχουμε κάποιον από την Επιτροπή εδώ που θα μπορούσε να μας επεξηγήσει κάπως ε, αυτή την κατάσταση. Ευχαριστούμε κυρία Φιγκερέδο, κυρία Μπάουερ. Με συγχωρείτε που παρεμβαίνω για άλλη μια φορά. Θα πρέπει να έχουμε κατά νου ότι θα πρέπει να δούμε πώς μπορούμε να βοηθήσουμε το Ινστιτούτο Ισότητας μεταξύ των δύο φύλων. Διότι δεν, έχουν, ε, δεν έχει επαρκές προσωπικό μιλά για πρόσληψη 9, μάλλον συγγνώμη, 6 ατόμων επί του χρόνου και αυτό που αναφέρθηκε είναι ότι από το Δεκέμβριο θα πρέπει να καταβάλουν ένα μίστομα. Και το μίστομα δεν είναι καθόλου ευκαταφρόνητο. Και νομίζω ότι θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μια αύξηση της χρηματοδότησης και όχι μείωση. Νομίζω λοιπόν ότι δεν θα μπορέσει να επιβιώσει το Ινστιτούτο αυτό. Νομίζω ότι θα πρέπει να δούμε ποιες είναι οι συνέπειες αυτής της κατάστασης και να παρέμβουμε δραστικά με την Κομισιόν διότι η κατάσταση είναι δραματική του Ινστιτούτου. Ευχαριστούμε πολύ κυρία Μπάουερ. Βλέπουμε ότι η κατάσταση θα πλήξει ιδιαίτερα το Ινστιτούτο Ισότητας ε, μεταξύ των δύο φύλων. Είναι τραγική κατάσταση. Δεν ξέρω κατά πόσο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να μας απαντήσει μερικώς. Εάν όχι, νομίζω ότι η κατάσταση είναι απαράδεκτη. Απαράδεκτη γιατί δεν ήρθε κανείς από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να απαντήσει. Νομίζω ότι θα πρέπει να πετήσουμε στο μέλλον να είναι παρούσα η Ευρωπαϊκή Επίτροπη σε τέτοιες ε, συζητήσεις, γιατί είναι μείζονο σημασία. Η κυρία Ματέρα έχει το λόγο. Μάλλον, κυρία Ματέρα, βλέπω ότι ε, έχετε την υποστήριξη όλων πολιτικών ομάδων, δηλαδή μπορούμε να ενώσουμε τις δυνάμεις μας για να επιλύσουμε αυτά τα θέματα ισότητας των δύο Κυρία Πρόεδρε, πράγματι, δυστυχώς δεν είναι παρούσα η Επιτροπή. Αυτό μας ανησυχεί ιδιαίτερα και είναι και έλλειψη ε, σεβασμού απέναντι μας. Άρα, ως η συγγήτρια αυτής της γνωμοδότησης, εγώ θα ζητήσω να παρευρίσκεται πάντα κάποιος από την Κομισιόν, δηλαδή ε, θα προωθήσω αυτά που μου είπατε, είναι απαράδεκτο να μειώνονται τα κονδύλια για το Ινστιτούτο, του Βίλνιους, να υπάρχει αυτή η δραστική περικοπή κατά ένα εκατομμύριο ευρώ τη στιγμή που έχουν να καταβάλουν και ενίκιο, πρέπει να προσληφθούν 7 ε, επιπρόσθετοι υπάλληλοι και πριν δεν σας μίλησα και για κάτι άλλο που θα πρέπει να μας απασχολήσει. Δεν έγινε αποδεκτό κανένα πολιτικό σχέδιο αυτής της Επιτροπής. Δηλαδή μας δώσανε βαθμό δέλτα. Στο σχολείο είναι πολύ κακός βαθμός. Και νομίζω, εάν συμφωνείτε, ότι θα πρέπει να επιστήσουμε την προσοχή μας σε ένα ή δύο προγράμματα, πιλωτικά προγράμματα, τα οποία θα επανεγγράψουμε έτσι ώστε να γίνουν αποδεκτά. Γιατί είναι σαν να ήμασταν στο σχολείο και να αποτύχαμε. Πήραμε δέλτα. Δεν νομίζω ότι τα πιλωτικά μας σχέδια δεν ήταν αποδεκτά, θέλω να πω, ως προς την ουσία τους. Δηλαδή, όπως μας είπε η κυρία Γκουρμάη, θα μπορούσαμε να υποβάλουμε τροπολογίες και αυτό θα είναι το μέσον για να καταπολεμήσουμε αυτή την κατάσταση, δηλαδή κηρύσουμε πόλεμο, τέλος. τις επόμενες ημέρες ή στο εγγύς μέλλον, όταν αυτή η Επιτροπή ε, επαναλάβει τις εργασίες της, ίσως θα μπορούσαμε να συνεργαστούμε με τους ε, πολιτικούς εκπροσώπους μας, να δούμε ποιες τροπολογίες μπορούμε να υποστηρίξουμε, γιατί εγώ στο σχολείο δεν πήρα ποτέ δέλτα και δεν θέλω να αρχίσω να παίρνω δέλτα εδώ στο Κοινοβούλιο. Η eh, κυρία Γκουρμάη. Απλώ θα ήθελα να σα ξεκαθαρίσω ότι η επιστολή αυτή θα πρέπει να πάει στη Διονρετνία τη εξηγεί ότι αυτό είναι απαράδεκτο και το ότι έχουμε τέτοια θέματα ε, του προπολογισμού ή άλλα ε, είναι απαράδεκτο. Άρα θα πρέπει να μα δοθούν εξηγήσει. Επίση, αν υπάρξει τέτοιου είδου ε, περικοπή, ε, αναρωτιέμαι τι είδους ε, διαβούλευση εννοούν. Ποιος το ζήτησε. Χρειάζεται εξήγηση του γιατί γίνεται αυτό. Άρα θα πρέπει και η Επίτροπος να δώσει και αυτή τη μάχη της για την ε, ισότητα. Επομένως, μείνουμε σταθεροί στη γραμμή μας, να την καλέσουμε τον Σεπτέμβριο και να το συζητήσουμε. Γιατί δεν κάνει αρκετά για την ισότητα. Έχει ευθύνη για το θέμα και συμφωνώ με τους προλύσαντες. Δεν θέλουμε το θάνατο αυτού του θεσμικού οργάνου. Εμείς δεν θα παραιτηθούμε από το να υποστηρίζουμε το θεσμικό όργανο. Ευχαριστώ κυρία Παπαδοπούλου, έχετε το λόγο. Θα ήθελα να προσθέσω αυτό που άκουγα το, το εξή. Πριν πολλή χρόνια, όταν είχε την Προεδρία της Ένωσης η Γερμανία, προώθησαν την ε, πρόταση της κάλυψης του προϋπολογισμού επί τη βάση των ε, σώτων των δύο φύλων. Οπότε το άλλο θέμα είναι το πώς θα πιεστεί η Ευρωπαϊκή Ένωση. Τώρα που πρέπει να αποφασίσει για τον προπολογισμό να πλαισιώσει αυτή την ιδέα του gender budgeting αυτού, τη σώτας των φύλων μέσα από τον προπολογισμό. Γιατί αν αυτό ισχύσει, εάν η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν καλύψει το θέμα με τον κοινωνικό προπολογισμό, πώς περιμένει να το κάνουν αυτό τα κράτη-μέλη του κοινωνικού προπολογισμού. Και νομίζω ότι με την ιδέα μου συμφωνούν οι πολιτικές ομάδες. Άρα να γίνει, αυτό προτεραιότητα ε, για τον προπολογισμό. Και αν το καταφέρουμε αυτό θα πετύχουμε αυτό που θέλουμε. Ευχαριστώ κυρία Παπαδοπούλου. Από ό,τι διαπιστώνω είμαστε προσταθερές στη γραμμή μας ακριβώς να δώσουν τη μάχη για την ε, ισότητα. Οπότε η κυρία Ματέρα, η, η εισηγήτρια, θα πρέπει να φροντίσει ακριβώς το πώς θα προωθήσουμε αυτή την πρόταση, να μην υπάρξει ενός είδους περικοπή. Θέλουμε να προχωρήσει αυτό το θεσμικό όργανο, να τα πάμε καλύτερα και όχι χειρότερα. 19 Ιουλίου το μεσημέρι τελειώνει η προθεσμία για την υποβολή των τροπολογιών. ...13 Αυγούστου... ...πρόκειται να έχουμε το οριστικό κείμενο... ...και επομένως συνάδελφοι... ...έτσι θα συνεχίσουμε τις προσπαθίες μας... Ακριβώ νομίζω ότι αν δεν κάνω λάθος όλες οι πολιτικές ομάδες συμφωνούν. Έχω μια ιδέα. Ίσως θα μπορούσα να έρθω σε επαφή σύντομα με τους πολιτικούς εκπροσώπους, διότι στις 19 ε, Ιουλίου είναι η προθεσμία για τις τροπολογίες, μετά ε, έχουμε τις διακοπές. Εγώ μπορώ να εργαστώ κατά τη διάρκεια των διακοπών, όμως οι βοηθοί μου δεν θα συμφωνήσουν. Εγώ δεν έχω πρόβλημα. Εν πάση περιπτώσει, τα καταγράφω όλα αυτά. Θα εργαστούμε πριν από την ε, λήξη της προθεσμίας, γιατί στις 30 Αυγούστου, όταν θα πρέπει να ψηφίσουμε, θα πρέπει να έχουμε ένα συμπαγές μέτωπο και να είμαστε σαφείς για την απαρχή των εργασιών, γιατί θα θέλαμε να είμαστε σε θέση μάχης. Γι' αυτό θα ήθελα λίγο μετά τη συνεδρία της Επιτροπής να το συζητήσουμε. Ευχαριστώ, Ευχαριστώ κυρία Ματέρα γιατί ε, σημειώνουμε την πρότασή σας και κλείνουμε τη συζήτηση αυτό του θέματος. Βεβαίως είναι ένα θέμα το οποίο θα ξανασυζητήσουμε σύντομα. Το επόμενο θέμα είναι μια γνωμοδότηση η οποία αναφέρεται στην Ευρωπαϊκή Διάσταση στον Αθλητισμό, σημείο 15, και η, η συγγήτρια είναι η κυρία Μίνσκιν. Ε, θα ήθελα να ακούσω την κυρία Σνίσχυν και να μας πει ε, τα σχόλιά της επί του θέματος. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ήμουν ε, υπεύθυνη ε, για το θέμα της, του ρόλου των γυναικών εις ε, τον αθλητισμό, μία γνωμοδότηση που καταρτήσαμε ε, για την Επιτροπή Πολιτισμού. Έχω συμμετάσχει σε πολλές συνεδριάσεις και συνέδρια επί του θέματος. Έχω συναντηθεί με εκπροσώπους των Υπουργείων και του Πολωνικού Υπουργείου Αθλητισμού της κοινωνίας των πολιτών και ε, έχω περί λάβει μόνο ορισμένα ε, ε, δηλώσεις επί του θέματος στην έκθεση και τα υπόλοιπα θα τα υποβάλλω σαν τροπολογίες. Όσον αφορά το ρόλο των γυναικών εις τον αθλητισμό, ναι μεν δεν είναι παρκώς εκπροσωπούμενες ακόμη και γι' αυτό και στα κράτη-μέλη πρέπει να κινητοποιηθούν όλοι οι ενδιαφερόμενοι κατά τρόπον ώστε ώστε να εγγυηθούν ίση ε, συμμετοχή των γυναικών στο χώρο αυτό και να προωθήσουν τη συμμετοχή τους στον ε, αθλητισμό. Αυτό που έχει σημασία για μας είναι η συμμετοχή των γυναικών στην διαχείριση των αθλητικών οργανώσεων και εδώ η κατάσταση είναι τραγική. Μόνο 11% γυναικών συμμετέχουν στη διοίκηση των αθλητικών ομίλων και υπάρχουν πάρα πολλές οργανώσεις που δεν έχουν καμία ε, ε, γυναίκα εκπρόσωπο στα διοικητικά συμβούλια, πράγμα το οποίο πρέπει να αλλάξει. Πρέπει να πούμε κατόπιν ερεύνης ότι η αύξηση του αριθμού των γυναικών στις, στις, στις που είναι εισηγμένες στο χρηματιστήριο βελτιώνει τις επιδόσεις των ομίλων αυτών γιατί οι γυναίκες έχουν μια ιδιαίτερη οπτική γωνία. Όταν λοιπόν έχουμε ε, και άντρες και γυναίκες στα διοικητικά συμβούλια παραδείγματος χάρη υπάρχει μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα και ε, ένα μεγάλο ποσοστό των γυναικών ε, ε, θα πρέπει να μπορέσει να φτάσει στο 20%. Αυτή ήταν τουλάχιστον μία δήλωση την οποία είχαμε επιζητήσει και δεν πλησιάζουμε το, το επίπεδο αυτό. Βέβαια μέχρι να επιτευχθεί ο ο στόχος τουλάχιστον το 2015, έχουμε τέσσερα χρόνια, άρα έχουμε κάποιο χρόνο για να μπορέσουμε να ανακτήσουμε το χαμένο έδαφος. Το άλλο θέμα είναι η παιδεία. Ε, πρέπει να έχουμε κατευθυντήριες γραμμές, πρέπει να μπορέσουμε να συνδυάσουμε ε, την ε, φυσική αγωγή με την αρχή της ισότητας των φύλων, να μπορέσουν οι γυναίκες, ε, οι αθλήτριες να έχουν μια επαγγελματική δραστηριότητα συνδυασμένη με την οικογενειακή τους κατάσταση, να εκπροσωπούνται επαξίως ή στην αγορά εργασίας και ε, ε, όσον αφορά την προβολή υπάρχει διαφορά ε, διότι η προβολή των γυναικών στα μέσα ενημέρωσης δεν μας ικανοποιεί και προτείνω διάφορες λύσεις επίσης όσον αφορά τα χρηματοοικονομικά ζητώ να υπάρξει χρηματοδότηση από το κοινωνικό ταμείο και από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης και να μπορέσει να υπάρξει ένα ειδικό πρόγραμμα ανταλλαγών για τις γυναίκες αθλήτριες και να υπάρξουν ταμεία τα οποία θα προωθήσουν την ισότητα στον ε, χώρο του αθλητισμού. Ε, περιμένω βέβαια τα περαιτέρω σχόλια τα οποία θα θέλετε να μου κάνετε. Ευχαριστώ, κυρία Σενίνσκιν. Τώρα η κυρία Λούνατσεκ έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ την εισηγήτρια για το σχέδιο το οποίο υποβάλλεται για όλα αυτά τα οποία είπατε, με τα οποία συμφωνούμε, διότι και εγώ υπήρξα αθλήτρια και έχω ασχοληθεί με την οργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων στη χώρα μου ε, και έχω υπάρξει αθλήτρια. Λοιπόν, ε, θα, θα προβώ και σε τροπολογίες, αλλά έχω μερικά σχόλια σχετικά με την ε, ε, με την ε, Επιτροπή Πολιτισμού θα έλεγα να ξανακοιτάξει κανείς το ψήφισμα του Κοινοβουλίου του 2002. Ε, ήταν ένα ψήφισμα σχετικά με με τις γυναίκες στον αθλητισμό πρόκειται για το ψήφισμα 2280 του 2002. Πέραν αυτού πρέπει να δούμε διάφορα θέματα. Πώς θα μπορέσουν να συμμετέχουν περισσότερες γυναίκες στην ηγεσία των αθλητικών οργανώσεων. Ε, διότι έχουμε διαπιστώσει και στις επιχειρήσεις και στους άλλους τομείς ότι αυτό είναι δύσκολο. Θα μπορούσαμε επίσης να αναφέρουμε ορισμένα θετικά παραδείγματα και κίνητρα τα οποία μπορούν να δοθούν για να προωθηθεί το θέμα αυτό. Τα δίκτυα γυναικών όπου μπορούν να λοστηριχτούν οι γυναίκες για να προχωρήσουν και να προωθηθούν είδα τις άλλες προτάσεις σας, λέτε όχι κάτω από 30% και για τα δύο φύλλα ναι μεν, αλλά θα πρέπει να αποβλέπουμε τουλάχιστον στο 40%. Νομίζω ότι ε, αυτό είναι το ελάχιστο επίπεδο, διότι διαφορετικά εάν θέσουμε τον πύχη ακόμη πιο χαμηλά δεν θα καταλήξουμε πουθενά. Ένα άλλο θέμα που βρίσκω πολύ σημαντικό είναι η ποιότητα της ε, φυσικής αγωγής που αναφέρατε και πώς θα υπάρξουν καλές πρακτικές, πώς θα μπορέσουν τα σχολεία και οι αθλητικοί όμιλοι να προωθήσουν ε, τον αθλητισμό στο γυναικείο φύλλο όταν μεγαλώνουν, διότι στην αρχή ε, τα παιδιά ε, ασκούνται σε διάφορα αθλήματα, αλλά μετά πολλά πράγματα αλλάζουν και αρχίζει να μειώνεται η συμμετοχή στον αθλητισμό. Και αυτό το βλέπουμε σε διάφορες αθλητικές οργανώσεις ενηλίκων. Σε ορισμένε περιπτώσεις οι γυναίκες επανέρχονται, αλλά καλό είναι να υπάρχει μία συνέχεια και συνεχής ενασχόληση των γυναικών ε, με τον αθλητισμό. Ή στην Αυστρία, στη Βιέννη την πόλη μου, οι δημόσιοι χώροι οι οποίοι ε, προσφέρονται για τους νέους ε, για αθλητισμό συνήθως καταλαμβάνονται ως επτοπλίστων από αγόρια που παίζουν ποδόσφαιρο, μπάσκετ και κάποια στιγμή θα πρέπει να μπορούν ε, και τα κορίτσια ε, ε, να αθληθούν. Άρα πρέπει να εξηγήσουμε και στα παιδιά, στα αγοράκια, ότι πρέπει να αφήσουν τη θέση τους ώρες-ώρες και στις ομάδες κοριτσιών. Ε, πέραν αυτών ζητάτε να υπάρξει η δυνατότητα για τις γυναίκες να συνδυάσουν την επαγγελματική με την αθλητική του ζωή. Αυτό θα πρέπει όμως να ισχύσει και για τους άντρες. Είναι πιο δύσκολα τα πράγματα για τις γυναίκες, αλλά υπάρχουν ε, γυναίκες ε, που έχουν παιδιά, που θέλουν να μείνουν στην οικογένειά τους και χρειάζονται στήριξη και από τους άντρες τους και θα έπρεπε αυτό να τονιστεί. Π.χ. επιπλέον ε, οι ορισμένες ευρωπαϊκές αρχές ε, ε, το fair play το οποίο μπορεί να καταπολεμήσει την ξενοφοβία τις διακρίσεις νομίζω ότι είναι επίσης ένα θέμα που θα έπρεπε να τονίσουμε όσον αφορά τις γυναίκες στα μέσα ενημέρωσης βεβαίως συνήθως και αυτό το έχω δει ε, το, ε, στη μου, στο δικό μου άθλημα που είναι το αλπικό σκι. Ε, ότι εάν κάπου κέρδισε μία γυναίκα και έχασε ένας αθλητής άντρα, βλέπετε στην επικεφαλίδα την επομένη της εφημερίδας να αναφέρεται γιατί έχασε ο άντρα. Και με μικρά γραμματάκια κάπου λέγεται ότι μία γυναίκα κέρδισε. Ε, θα πρέπει λοιπόν ίσως να προβάλλουμε περισσότερο τις θέσεις των γυναικών. Και ε, να κοιτάξουμε και τα ε, κορίτσια των μεταναστών ε, διότι αυτές ίσως λόγω οικογενειακών καταβολών δεν επιτρέπεται να συμμετάσχουν σε αθλήματα όπως η κολύμβηση και θα πρέπει να προωθήσουμε και τη φυσική αγωγή και τον αθλητισμό να μάθουν να χρησιμοποιούν το σώμα τους θετικά και αυτά είχα να σας πω. Θα σας υποβάλω τις σχετικές τροπολογίες. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Λούνατσα και κυρία Φιγκερέντο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Όλα προελέχθησαν, με τα οποία συμφωνώ ως επιτοπλίστων. Θα ήθελα να ασχοληθούμε όμως με τις διακρίσεις που υπάρχουν, ιδιαίτερα ως προς τις γυναίκες αθλήτριες. Διότι αυτό το βλέπω και στη χώρα μου. Δηλαδή, όταν πρόκειται για απονομές, δεν υπάρχει ίδια αντιμετώπιση ανδρών και γυναικών. Και μπορώ να πω ότι πέρα από το θέμα της επικοινωνίας, των κοινωνικών διακρίσεων, των διακρίσεων γενικότερα ως προς τις επιδόσεις των γυναικών, βλέπω ότι και σε επίπεδο απονομής υπάρχει μία διαφορετική στάση. Αυτό το είχαμε αναφέρει και στο ψήφισμά μας, ένα ψήφισμά μας, ένα παλιό ψήφισμα του 2002. Θα πρέπει να δούμε τι μπορεί να κάνει η Κομισιόν επί του θέματος, δηλαδή ποιες είναι οι χρηστές πρακτικές και ούτω καθεξής. θα μπορούσαμε να βρούμε κάποιο τρόπο για να καταπολεμήσουμε αυτό το, αυτά τα επίπεδα διακρίσεων. Βεβαίως θα πρέπει να υπάρχουν κίνητρα για τον αθλητισμό και τα κίνητρα αυτά δίνονται ήδη από το σχολείο, όταν τα παιδιά είναι μικρά. Θα πρέπει λοιπόν ε, να υπάρχει ένα μεγάλο κίνητρο για τα νέα κορίτσια, για τα μικρά κορίτσια. Για να καταπολεμήσουμε αυτή τη ε, διάκριση που υπάρχει ως προς την δύσκολη προσπελασιμότητα των γυναικών στο χώρο του αθλητισμού. Εάν δεν προωθούμε τον αθλητισμό ήδη από τα παιδικά χρόνια, δεν θα σταματήσει αυτή η γενικότερη διάκριση σε επίπεδο κοινωνίας. Θα πρέπει λοιπόν να δίνουμε όλο ένα και μεγαλύτερη προσοχή στον αθλητισμό για τα ε, μικρά κορίτσια, για, τα, για τις γυναίκες που αρχίζει, κάτι το οποίο αρχίζει από τη δημόσια εκπαίδευση, από τα ε, χρόνια ήδη του δημοτικού και δεν μιλάω για αθλητισμό, για ελιτίστικο αθλητισμό, αλλά αθλητισμό για όλους τους πολίτες. Θα υποβάλουμε και ορισμένες προτάσεις προς την εισηγητριά μας. Και ελπίζω να λάβει υπόψη και τις δικές μου προτάσεις. Ο κύριος Ταραμπέλα. Merci, Madame la Présidente. Je voulais saluer la euh, Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε και για αυτή την έκθεση που είναι τόσο σημαντική. Γιατί ε, είναι πάρα πολύ σημαντική υπόθεση ο αθλητισμός και χθε δεν άκουσα την κυρία Ζαμπόσκα για την ε, ε, εγκληματικότητα των νέων και λοιπόν νομίζω ότι θα πρέπει να συνδέσουμε το πρόβλημα αυτό των ε, νέων εγκληματιών με τον αθλητισμό και ακριβώς να αναδείξουμε το ότι ο αθλητισμός θα πρέπει να προθεθεί για τους ε, νέους και ότι θα πρέπει οι νέοι να ξεκολλήσουν από τα παιχνίδια στους κομπιούτερ και είναι το πνεύμα της ομαδικότητας, είναι μια αλληλεγγύη όταν ε, όταν τον, τον, τον παίζουν λοιπόν σε ομάδες μπάσκετ, ή ποδόσφαιρο ας πούμε κάποιος συμπέκτη όταν αρρωστήσει, προσπαθεί να πάει να αφήσει έτσι την ομάδα και το ποδόσφαιρο επομένω και το μπάσκετ. Ε, ο σεβασμός προς το διαιτητή, ε, όπως άλλωστε γίνεται κυρίως ε, από τους Αγγλοσάξονες και βεβαίως ότι ακριβώς μαθαίνουν ότι υπάρχουν κάποια κάποια όρια που δεν πρέπει κανεί να υπερβεί, επομένως να ποια είναι η εκπαιδευτική αξία του, του, του, του, του σπόρου του αθλητισμού. Έχουμε άλλωστε και το παγκόσμιο ε, κύπελο. Ε, η Σουηδία αποκλείστηκε, η Παγκοσμίου των Γυναικών και η Γαλλία. Κρίμα για τη Σουηδία, κρίμα και για τη Γαλλία. Αποκλείστηκαν νωρί. Όμω ε, η, Γερμανία που πρέπει να αναγνωρίσουμε έχει αυτό το, το, το, καλό ότι αναδεικνύει το γεγονό. Όμω δεν το ανέδειξαν το ίδιο, δεν το προέβαλαν και άλλε χώρε. Και άρα θα έπρεπε να. Ε, να προβάλλεται όπως γίνεται και με ε, τα μάτς των ε, ανδρών ε, που ξέρουν πολύ καλά πόσο, πόσο τα, τα τηλεόραση και μου ότι θα πρέπει να ξεπεραστεί και αυτό το στερεότυπο. Επίσης θα ήθελα να σταθώ στον ρόλο των αθλητών υψηλού επίπεδου, ο, ο Μπιόρν Να είδατε όλα έχουν κολλήσει με στη Σουηδία σήμερα, δεν ξέρω γιατί. Και ο Μπιόρν Μπόργ έλεγα ότι δίνει το παράδειγμα είχε πάρει αντί για ρακέτα του πινκ-πονγκ, ήταν τα 14, πήρε μια ρακέτα ε, του τέννις και είδατε που έφτασε, οπότε υπάρχουν άλλωστε και χιλιάδες ε, μετά που τον ακολούθησαν στη Σουηδία και έχουν την Kim Kleister ε, στο Βέλγιο, που επομένως το τέννις ξέρουμε ότι προβάλλεται πολύ από τα ΜΜΕ ε, υπάρχουν όμω και άλλα σπορτα, τα οποία προβάλλονται λιγότερο, οπότε θα πρέπει καθ' αυτόν τον τρόπο να προβάλλονται οι αθλητέ και οι πιο ανώνυμοι. Αλλά όμω και αυτόν ο ρόλο είναι ε, εκπαιδευτικό, είναι παραδείγματα προ μίμηση. Και για αυτόν τον τρόπο οι νεότερε γενιέ ε, ελκύονται και προσπαθούν να ακολουθήσουν το παράδειγμα αυτών των αθλητών. Και επίση, κατακλείδη να σα πω για το σημείο 8, ότι συμφωνώ ότι θα πρέπει να κληθεί η Κομισιόν και τα κρατημέλη να συγχρηματοδοτήσουν κάποιε υποδομέ που να είναι για τι ανάγκε των γυναικών. Και προσοχή, ε, θα ήθελα να σα πω ότι ε, έχουμε αυτού του είδους ε, που λέμε θα πρέπει να είναι χωριστά για λόγους θρησκευτικού κοριτσάκια από αγορά και τον καταθλιτισμό. Αυτό εγώ δεν το βρίσκω σωστό. Ε, ε, ξέρετε και τώρα που έχουμε την κρίση θα πρέπει να κάνουμε προσπάθεια ε, να εξοικονομούμε χρήματα. Επομένως είναι σπατάλη χρημάτων το να έχουμε δύο πισίνες, μία για αγορά και μία για κοριτσάκια. Ευχαριστούμε κύριε Ταραμπέλα, λέει η πρόεδρος. Και τώρα δώσω το λόγο στην κυρία Στρέλα, θα ήθελα και εγώ να σας πω τις παρατηρήσεις μου πρώτα-πρώτα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Ταραμπέλα ε, που αναδείξατε τις ε, χθεσινές προσπάθειες των ε, Σουηδών, των Σουηδέζων μάλλον. Κρίμα, κρίμα, δεν περάσαμε στο τελικό. Και θα ήθελα επίσης να σας πω και κάτι άλλο για τη συζήτησή μας. Πολύ σωστά είπατε ότι ο αθλητισμός ενώνει και θα πρέπει ακριβώς να αναδειχθεί ο εκπαιδευτικός ρόλος των σπορ και το πόσο είναι οι αθλητές παραδείγματα προς μίμηση. Συμφωνώ με αυτό που είπε και η κυρία Λούνατσικ προηγουμένως. Με εντυπωσιάσατε με αυτό που είπατε. και βλέπουμε πόσο ε, ε, αρέσει ο αθλητισμός στα παιδιά και επίσης να αναδειχθεί το γεγονός ότι με τον αθλητισμό εάν κάποια κοπέλα ασχολείται ε, αυτό την προστατεύει και επίσης δεν θα πρέπει ε, να έχουν παθητικό ρόλο οι κοπέλες και όταν ας πούμε φτάνουν στην εφηβεία να σταματάνε τον αθλητισμό, απλά παθητικά να βλέπουν τους ε, άντρες, τους, τα παλικαράκια που αθλούνται, επομένως θα πρέπει να συνεχίσετε ο αθλητισμός και, και, και από την εφηβεία και μετά. Μην συνεχίζουν μόνο τα αγόρια Βεβαίω και καμιά φορά είναι πιο δύσκολο για τι κοπέλε να συνεχίζουν το σπορ, αλλά παρουσιάζει ενδιαφέρον το θέμα. Θα πρέπει να το βάλουμε στο σωστό πλαίσιο, να το εξετάσουμε, να το μελετήσουμε πολλέ φορέ. Ε, ε, πολλές φορές υπάρχει ένας, ένας ελιτισμός που πρέπει ανέβει και στον αθλητισμό και, και αυτό ελκύει περισσότερο τα αγόρια παρά τα κορίτσια. Άρα θα πρέπει και τα κορίτσια να συνεχίζουν αυτόν τον δυναμικό ρόλο του, που, που έχει το σπορ ε, και γενικά έχουν δυναμισμό στην κοινωνία και εμείς επομένως έχουμε την, ε, το καθήκον να φωτίσουμε αυτές τις πτυχές του θέματος και σε ορισμένε ε, χώρες βλέπουμε πώς λειτουργεί η υπόθεση σαν παράδειγμα και ε, επίσης θα πρέπει θα πρέπει τα αθλητικά γεγονότα που συμμετέχουν γυναίκες να προβάλλονται, να προβάλλονται σε ώρα υψηλή τηλεθέασης, όπως γίνεται και με τους άντρες. Επίσης, τα σπορ των γυναικών ε, θα πρέπει και αυτά να γίνονται με οργάνωση όπως γίνεται και με τους άντρες, με συλλόγους, με διεθνείς ομοσπονδίες Επίσης ε, υπάρχει, υπάρχουν κάποιοι περιορισμοί, όπως ας πούμε ότι η Ομοσπονδία Τέννης Γυναικών έχει επιβάλει να παίζουν με φουστίτσες οι κοπέλες το οποίο είναι γελίο. Επίσης ε, και ο ποσφαίρο γυναικών υπάρχουν αντίστοιχοι περιορισμοί, ε, ειδικά ρούχα, ειδικοί χώροι. Μα δεν είναι δυνατόν να θεωρήσουμε ότι οι αθλήτριες είναι φιλικά αντικείμενα που αθλούνται. Όλα αυτά έχουμε ευθύνη να τα αναδείξουμε. Δεν, θέλουμε να, να, να, να υπάρχει τέτοια αντιμετώπιση, τέτοιες προκαταλήψεις για τις ε, αθλήτριες. Κυρία Εστέλα, ε, συμφωνώ με όσα ελέγχθησαν και θα ήθελα να συγχαρώ την εισηγήτρια, εξαιρετική εργασία της. Θα ήθελα να τονίσω τρία στοιχεία. Το πρώτο σχετίζεται με την ε, άσκηση καθαρά, ανεξάρτητα δηλαδή από την ηλικία, το φύλλο, ο άνθρωπος πρέπει να κινείται πέρα δηλαδή από κοινωνικο-οικονομικούς παράγοντες, θα πρέπει κανείς να αθλείται. Το δεύτερο ζήτημα έχει σχέση με τους αθλητές υψηλών επιδόσεων και εδώ μιλώ για τις αθλήτριες. Είδαμε ότι ακόμα και οι γυναίκες Ολυμπιονίκες έχουν πρόβλημα να επανέλθουν στην, ε, στη φυσική τους δραστηριότητα μετά από ένα μετάλλιο. Δηλαδή, πολλές φορές υπάρχει μια στασιμότητα μετά. Νομίζω λοιπόν ότι για τους νεότερους θα πρέπει να γίνει μια μεγάλη εργασία με τα σχολεία έτσι ώστε να δώσουμε κίνητρα για τους νέους ως προς, την, ε, ως προς τον αθλητισμό. Συμφωνώ με αυτά που είπε η κυρία Φιγκερέλο ως προς την απονομή μεταλλίων. Θα ήθελα να πω ότι αυτό που συμβαίνει με την απονομή είναι αυτό που συμβαίνει με τους μισθούς. Δηλαδή οι γυναίκες για την ίδια εργασία λαμβάνουν 18% λιγότερο. Το ίδιο ισχύει και με τα έπαθλα που έχουν άλλο αντίκτυπο για τις γυναίκες σε σχέση με τους άνδρες. Αυτό <coughs> μπορεί να αλλάξει. Θα σας πω ότι έγινε με μένα όταν ήμουν δήμαρχος της Σύντρα και είχαμε προωθήσει αθλητικές δραστηριότητες. Όταν είχαμε την αρχική πρόταση για την χρηματοδοτική υποστήριξη, ήθελα εγώ να δω τον κανονισμό και είδα ότι για τις γυναίκες το έπαθλο, δηλαδή το συνολικό ποσό ήταν κάτι λιγότερο από το ίμιση σε σχέση με τους άνδρες και είπα ότι εγώ δεν μπορώ να δεχτώ τη διοργάνωση διότι εδώ πρόκειται για διάκριση των αθλητριών. Αυτό δημιούργησε μεγάλη αναταρχή. αλλά ε, και επειδή ακριβώς έπρεπε να αναλάβουμε τη διοργάνωση, άλλαξε ο κανονισμός. Ήταν η πρώτη φορά που φάνηκε το όνομά μου στο ίντερνετ, διότι οι αθλήτριες βάλαν τη φωτογραφία μου με αυτή την απόφαση που θεωρούσαν παραδειγματική. Δηλαδή, πολλές φορές με συγκεκριμένες χειρονομίες ή θέσεις ο καθένας στο επίπεδό του μπορεί να οδηγήσει σε μία διαφοροποίηση και να αλλάξουν καταστάσεις. Θα μπορούσαμε να πούμε στην Επιτροπή ότι δεν πρέπει να δέχεται κανονισμούς που αποτελούν διάκριση για τις γυναίκες. Είναι παράδεκτο αυτό. Και αντιτίθεται σε αυτό που προβάλλουν ε, οι ίδιες οι συνθήκες. Αυτή είναι η δική μου εμπειρία, έτσι τα έζησα εγώ τα πράγματα και ε, το αποτέλεσμα ήταν άκρος θετικό. Ευχαριστούμε κυρία Στρέλα Δίνουμε το λόγο στην Επιτροπή τώρα. Έχετε το λόγο. Sorry, on this side. Συγγνώμη που κάθομαι από αυτή την πλευρά. Apologies for, for my seating here. Thank, thank you very much. I think it... Σας ευχαριστώ. Είδα την ανακοίνωση για τον αθλητισμό όπου λέμε ότι θα προωθήσουμε ε, διασυνοριακά projects έτσι ώστε οι γυναίκες να βρίσκονται σε καλύτερη θέση Νομίζω λοιπόν ότι θα συμπεριλάβουμε και όλες τις άλλες πτυχές που αναφέρατε, γιατί είναι μεγάλο πρόβλημα για τον αθλητισμό και η κυρία Βασιλείου ήδη εξέφρασε πολλές φορές την άποψή της ότι θα πρέπει οι κυβερνήσεις να είναι κοινωνεί σε όλες τις αθλητικές, αθλητικές δραστηριότητες και το ίδιο θα κάνει και στην Επιτροπή ε, Γυναικών στον Αθλητισμό που θα συνέλθει στο Λονδίνο το Σεπτέμβριο. Την προηγούμενη εβδομάδα ο αθλητισμός συμπεριελήφθη σε μία ε, πρώτας Επιτροπής, δηλαδή στο πολιετές πλαίσιο. Άρα ο αθλητισμός θα συμπεριλαμβάνεται σε αυτό το νέο χρηματοοικονομικό πλαίσιο και στις ε, δημοσιονομικές πρόπτικες και τότε θα μπορέσουμε να υλοποιήσουμε αρκετές από αυτές τις πτυχές. Η Επιτροπή κρίνει ότι θα πρέπει να συνεργαστούμε με το κίνημα του αθλητισμού που είναι αυτόνομο βεβαίως, αλλά συζητώντας από κοινού θέματα θα φτάσουμε σε αυτά αποτελέσματα. Ε, επίσης, αξιολογούμε διάφορα σχέδια που έχουμε μέσα στα πλαίσια των προπαρασκευαστικών δράσεων και η Επιτροπή σας θα πρέπει να τονίσει τα αποτελέσματα του σχεδίου Ολύμπια όπου έχει χαρτογραφηθεί η ισότητα των δύο φίλων στον αθλητισμό. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Και επίσης θέλω να σας πω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικά όσα είπατε και θα λάβω υπόψη ό,τι έχετε πει. Ευχαριστούμε, κυρία εισηγήτρια. Για τις τροπολογίες τώρα. 29 Αυγούστου εκπνέει η προθεσμία υποβολής των τροπολογιών και θα συζητηθεί εδώ στην Επιτροπή μας στις 15 Αυγούστου και 5 Οκτωβρίου στην κυρία Σορμοδία Επιτροπή. Τώρα πάμε στο επόμενο σημείο της διατάξεως, το σημείο 16. 16 που αφορά τις μόνες γυναίκες, τις γυναίκες που μεγαλώνουν μόνες τα παιδιά τους. Κυρία Ματέρα. Και στο παρελθόν ε, είχαμε συζητήσει υποτύπων ε, προετοιμασία το ίδιο θέμα στην Επιτροπή μας. Τώρα θα πρέπει να δούμε τις τροπολογίες οι οποίες έχουν υποβληθεί. Έχετε το λόγο κυρία Ματέρα. Grazie Presidente. Allora, eh, ringrazio tutti i colleghi per aver... να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους που συνεργάστηκαν για την έκθεση αυτή έχουμε 164 τροπολογίες. Ήθελα να ευχαριστήσω τους σκιώδεις που συνεισέφεραν και εκείνοι και ήταν διαθέσιμοι μέσα σε διμερείς συνεννοήσεις, στα πλαίσια διμερών συνεννοήσεων. Το θέμα είναι αρκετά σαφές. Έχουμε 11 τροπολογίες συμβιβασμού και θα ήθελα να υπενθυμίσω στους συναδέλφους ότι στις 15 Σεπτεμβρίου θα ψηφίσουμε στο Στρασβούργο. Τώρα, εργαζόμενοι για τις ε, τροπολογίες προσπάθησα να σταθώ στα συγκεκριμένα μέτρα για τις μητέρες που μεγαλώνουν τα παιδιά τους μόνες. Δηλαδή να προβάλλω μία έκθεση συνεκτική αλλά και με πολλά επιμέρους θέματα και συγκεκριμένα μέτρα. Γι' αυτό Γι' αυτό και έκοψα τις τροπολογίες που ήταν εκτός θέματος, ας το πούμε έτσι. Έπρεπε να λάβω υπόψη το γεγονός ότι ορισμένες ε, καλές τροπολογίες μιλούσαν και για μονογονικές οικογένειες όπου μεγαλώνει το παιδί ο πατέρας. Ήδη είχαμε μία συζήτηση την προηγούμενη φορά και εσείς ήσασταν αρκετά αποφασισμένοι να ακολουθήσετε το βασικό θέμα το οποίο εμπεριέχεται και στον τίτλο, δηλαδή τις μόνες, τις μητέρες, ε, τις, μόνες, τις μητέρες μεγαλώνουν μόνο στα παιδιά τους. Άρα, ε, ίσως στο μέλλον θα μπορούσαμε να έχουμε ε, τροπολογίες και για single fathers και όχι μόνο single mothers. Δηλαδή να δούμε τις ε, μονογονεϊκές οικογένειες στο μέλλον χωρίς να προσδιορίζουμε το φύλλο του γονέα. Επειδή λοιπόν θα πρέπει να υπάρχει σαφήνεια και διαφάνεια και θα πρέπει να είμαστε και αρκετά συνεκτικοί ε, βρίσκοντας καλές λύσεις δεν θα λάβω υπόψη τις τροπολογίες όπου γίνεται λόγος για πρόληψη διότι πρόκειται για μία έκθεση που αντιμετωπίζει το πρόβλημα δίνοντας λύσεις δεν μιλάμε μόνο για την πρόληψη που είναι σημαντική, γιατί μιλάμε για τη χρήση αντισύλληψης ή τα μέτρα για την αποφυγή του διαζυγίου. Μιλούσα λοιπόν για συγκεκριμένη αρρωγή προς τις ε, μητέρες που μεγαλώνουν μόνες τα παιδιά τους. Το είδα λοιπόν το θέμα αυτό και με άλλες ε, πολιτικές ομάδες. Έχει μεγάλη σημασία να υπάρχει και η σωστή εκπαίδευση. Για να δούμε πώς ε, ε, γίνεται η επαφή και με το άλλο φύλλο, δηλαδή να υπάρχει μία εκπαιδευτική διάσταση ήδη από το σχολείο. Σας υπενθυμίζω ότι μιλάμε για ένα μεταβατικό ας πούμε θέμα. Αυτός είναι ο κύκλος της ζωής βεβαίως. Ελπίζουμε όμως ότι οι μητέρες δεν θα είναι μόνες, διότι θα βρουν ένα νέο σύντροφο και θα δημιουργήσουν ένα νέο οικογενειακό πυρήνα. Αυτό έχει μεγάλη σημασία και γι' αυτό μιλάμε για μεταβατικά μέτρα, δηλαδή προσωρινά. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ κυρία Ματέρα ή κυρία Γκουρμάη. Κυρία Γκουρμάη θέλετε να παρέμβετε. Ευχαριστώ. Ε, βέβαια πρέπει να υπάρχει ίση μεταχείριση. Λοιπόν, Καταρχήν θέλω να ευχαριστήσω την εισηγήτριά μας για την εργασία της και βεβαίως πιστεύω ότι αυτή η έκθεση δείχνει τι δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι ε, ε, γυναίκες που μεγαλώνουν τα παιδιά τους μόνες τους. Ε, η κατάσταση αυτή στην Ευρώπη δεν είναι μια εξαίρεση γιατί ξέρουμε ότι παρουσιάζεται παντού τα τελευταία χρόνια. Δεν θέλω όμως ε, οι οικογένειες αυτές να μείνουν αποκλεισμένες από τα ωφέλη και θεωρώ ότι ε, και μια γυναίκα με το παιδί της αποτελούν μια οικογένεια και πολλοί από εμά γνωρίζουν πόσο δύσκολο είναι να συνδυάσει κανείς την επαγγελματική επαγγελματική ζωή με την ε, ε, ιδιωτική. Εάν λοιπόν ε, οι οικογένειες ε, ε, αντιμετωπίζουν προβλήματα, αντιλαμβάνεστε πόσο πιο δύσκολη είναι η κατάσταση όταν είναι μονογονικές οικογένειες όπου υπάρχει μεγαλύτερη δυσκολία προσβάσεως στην αγορά εργασίας, οικονομικά προβλήματα τα οποία συνδυάζονται και ένα, μια διαφορά ως προς τις συντάξεις. Ε, πρέπει λοιπόν κανείς να αντιληφθεί ότι πλέον, πλέον των διακρίσεων υπάρχουν ε, και άλλοι παράγοντες ε, όπως οι ανεύθυνες μητέρες ε, υπάρχει μία διάκριση η οποία θα πρέπει να καταργηθεί, να διευκολύνουμε ε, την ε, ζωή των γυναικών που μεγαλώνουν τα παιδιά τους μόνες τους και όπως ανέφερα η έκθεση αποτελεί μια καλή βάση διότι επιτρέπει να δούμε ποια είναι η βάση της εργασίας μας και εν ονόματι της πολιτικής μου ομάδος ε, ήθελα να σας πω ότι θα την υπερψηφίσω αλλά θέλω να αναφερθώ και σε ορισμένα επιπλέον θέματα τα οποία θέλουμε να περιλάβουμε εις ε, τις τροπολογίες μας ε, όσον αφορά την ε, δυνατότητα περιθάλψεως των παιδιών σε καλές τιμές, αξιόπιστες, σοβαρές και μόνο έτσι θα μπορέσουν οι γυναίκες να συνεχίσουν την εργασία τους ή τη σπουδές τους. Δεν χρειάζεται οι γυναίκες να εγκαταλείψουν το παιδί τους για να ε, ε, δραστηριοποιηθούν επαγγελματικά. Πρέπει λοιπόν να υπάρξει περίθαλψη των παιδιών. Χρειάζεται επίσης η δυνατότητα να βοηθήσει τις μητέρες αυτές να δραστηριοποιηθούν και να γίνουν αξιόπιστα μέλη της κοινωνίας. Και γι' αυτό θα πρέπει να υπάρξουν κίνητρα που θα προωθήσουν αυτές τις ρυθμίσεις και ο καθένας θα, ξέρει, θα πρέπει να ξέρει ε, τι πρέπει να αναλαμβάνει ο καθένας. Είμαστε βέβαια σε μια περίοδο οικονομικής κρίσεως και αυτό διευκολύνει να επιβαρύνει κανείς τις γυναίκες και γι' αυτό πρέπει να φροντίσουμε ε, να μπορούν οι γυναίκες και ιδίω ε, οι γυναίκες που μεγαλώνουν μόνες τους τα παιδιά τους να ενισχυθούν ε, για να μπορεί να υπάρξει βοήθεια πριν η τεκνοποίηση γυναίκα στη συνέχεια ε, και στο τέλος η σύνταξή της ε, μπορεί να είναι πολύ χαμηλή ε, διότι δεν είχε ποιοτική εργασία την εποχή που μπορούσε να είναι δραστήρια για να φροντίσει μόνη της το παιδί της. Είναι ένας φαύλος κύκλος τον οποίον ήδη ανέφερα και γι' αυτό η ε, συγητριά μας η Μπάρβαρα προσπαθεί να μας παρουσιάσει το θέμα και ελπίζω ότι θα μπορέσουμε να ψηφίσουμε την έκθεση αυτή πολύ, με μια πολύ καλή μορφή και ε, θα συμβάλλω σε, σε συμβιβαστικές τροπολογίες. Η κυρία Στρέλα έχει τώρα το λόγο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε και εγώ να συγχαρώ την εισηγήτρια που πήγε πάρα πολύ καλά. Eh, τώρα θα πρέπει να δούμε τι θα γίνει με τις τροπολογίες. Ε, διότι είχα υποβάλει κάποιες τροπολογίες που δεν τις δέχθη η συγγήτρια. Και αυτό το οποίο ήθελα ήταν να ζητήσουμε η ίδια δικαιώματα για όλους τους γονείς και για τους γονείς που μεγαλώνουν μόνοι τα παιδιά τους. Φεμινιστικά το βλέπω. Θα πρέπει επίσης ε, να είμαστε συνεπείς σε αυτά που ζητούμε και θα πρέπει επίσης με συνέπεια να καταπολεμούμε κάθε δυσμενή διάκριση. Για μένα και η πατρότητα και η μητρότητα είναι ε, δύο όψεις του ίδιου νομίσματος. όπως κάνουμε και με την ε, άδεια μητρότητος, που ζητήθηκε και θεσπίστηκε και η άδεια πατρότητος. Οπότε, Ακριβώ όπως θέλουμε να κατακτήσουμε κάποια δικαιώματα για τις μητέρες γονεμόνες στα παιδιά τους και θα πρέπει να είμαστε συνεπείς και να ζητήσουμε ακριβώς η διαρρύθμιση και για τους πατέρες που μεγαλώνουν μόνοι τα παιδιά του. Οι μονογονεϊκές οικογένειε, δηλαδή. Υπάρχουν και μονογονικές οικογένειες που αποτελούνται από πατέρα και παιδιά. Ποιε είναι οι εξαιρέσει σχέση με τις μητέρες μεγαλών τα παιδιά. Οπότε, ε, παρακαλώ θα πρέπει να ε, δεχθεί η συγκεκριμένη την τροπολογία μου. Αλλιώ, νομίζω ότι δεν θα είμαστε συνεπεί σε αυτά που πρεσβεύουμε. Ακριβώς επειδή πάντοτε θέλουμε να ισχύουν οι ρυθμίσει για τις και γυναίκε ε, σε αυτό το επίπεδο, όπω και για τι άδειε, και επίση το ίδιο να γίνει ε, όπως είχαμε πει και ε, να, να, να, μην, να μην θεωρείται η γυναίκα αντικείμενο. θέλουμε τα στερεότυπα, θέλουμε οι ερμηνείς διακρίσεις να καταπολεμούνται. Ο πατέρα, επομένω φυσικά ε, θα πρέπει και αυτός να θεωρείται μόνο οικογένεια να μόνο στα παιδιά. Επότε θα παρακαλώ να το λάβει αυτό υπόψη η συγκεντρία. Και ε, δεν νομίζω ότι εάν βάλουμε τη ρύθμιση αυτή που ζήτησα στην οδηγία, δεν νομίζω ότι θα είναι αυτή η ρύθμιση εκτός θέματος, εκτός του πεδίου ε, του, του, του πελληνικούς αυτής της ε, ε, εκθέσεως. Να είμαστε επομένω συνεπείς να καταπολεμούμε πάσα δυσμενή διάκριση. Η Πρόεδρος. Κυρία Στρέλλα, σας ευχαριστούμε. Κύριε Παρβανόβα. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ και εγώ να ευχαριστώ την, την εισηγήτρια, την κυρία Ματέρα, για την εκθεσή της, για όλα αυτά τα οποία μας απασχόλησαν, που συζητήσαμε σύμφωνα με την προσέγγιση της και θα καταλήξουμε τελικά στην κεντρική εκδοχή αυτή την ε, έκθεση και στους συντονιστές τους κάναμε λάθος που είπαμε ότι θα κάνουμε έκθεση μόνο για τις μητέρες με τον τα παιδιά τους και θα έπρεπε να είμαστε πιο ευέλικτοι για να καλύψουμε και τους άνδρες. Οπότε, τουλάχιστον στην τελική έκθεση, να φύγει το ζήτημα των ε, πατέρων μεγάλων μόνοι τα παιδιά. Και αυτό επομένω θα πρέπει να το λάβουμε υπόψη για τη δουλειά μα στο μέλλον. Και ενδεχομένω να κάνουμε μια ολόκληρη έκθεση για του πατέρε μεγάλων μόνοι τα παιδιά, ε, α πούμε του χρόνου. Επίση, κάτι άλλο. Όταν μιλούμε για αυτέ τι μητέρε, μόνε, ε, μην παρά αυτά που ελέγχθησαν για την οικονομική διάσταση του θέματος και για τις ρυθμίσεις του κάθε κράτους μέλους, αλλά θέλω να σταθούμε στο πόσο σημαντικό είναι, θα πρέπει να αναδείξουμε δηλαδή ότι να, ενθαρρυνθούν τα ε, κράτη-μέλη να συνεργαστούν με το Ίδρυμα Ισότητας. Και θα πρέπει επομένω η μία χώρα μετά την άλλη να δώσει κάποια στοιχεία, να συγκριθούν αυτά τα στοιχεία, να δούμε ποιε είναι οι άριστε πρακτικέ είναι σημαντικό και κατά αυτόν τον τρόπο νομίζω θα αποκτήσει νέα διάσταση το έργο του Ινστιτούτου Ισότητας. Υπάρχει εδώ πέρα θέμα το οποίο δεν έχουμε ασχοληθεί ακόμα. Υπάρχει και ενώ επίσης θα πρέπει στην έκθεση να μην παραλείψουμε, να αναφέρουμε ότι πρέπει να καλύψουμε και τις γυναίκες που είναι έγκυες και τις γυναίκες που μετά γεννούν τα παιδιά αλλά και θα πρέπει μέσω ε, σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης να δουλέψουμε και πάνω στο θέμα των επιθυμήτων ε, ε, εκείσεων. Οπότε, να δούμε μέσα από κοινότητες, από όλους τους φορείς τι γίνεται με τις εγκυμοσύνες πριν τα 18 Βέβαια, πολλές φορές το δίκαιο το απαγορεύει. Όμως, έτσι κι αλλιώς σε κάποιες κοινωνίες, σε κάποια μέρη ε, συμβαίνει αυτό συχνά. Παρά λοιπόν το, ότι ισχύει πέρα του αντιθέτου νομοθεσία. Αυτά ήθελα να σας πω. Ελπίζω ότι θα έχουμε τον χρόνο για να συζητήσουμε ξανά την έκθεση στο μέλλον και επί τη βάση της ε, αγαστής συνεργασίας που ήδη έχουμε. Ευχαριστούμε κύριε Παρβάνοβα. Κύριε Μπιλμπάου. Ευχαριστώ πρόεδρε. Για να μην επαναλάβω πράγματα που προελέχθησαν, θα ήθελα να μιλήσω μόνο για τις δικές μας τροπολογίες. Καταρχήν, νομίζω ότι η κακή εικόνα που υπάρχει για τις ανήπαντερες μητέρες μπορεί να αλλάξει στα κράτη-μέλη. Υπάρχουν πολλές ευρωπαϊκές χώρες και περιφέρειες που έχουν ένα πολύ καλό ρυθμιστικό πλαίσιο και δεν ζουν οι μητέρες κατά αυτόν τον τρόπο. Έχουμε υποβάλει τροπολογίες και νομίζω ότι μπορούμε να δούμε τις αντιδράσεις των γυναικών ήδη σήμερα, γιατί τη στιγμή που υπάρχει οικονομική ανάπτυξη υπάρχουν πολλές γυναίκες που επιλέγουν το να ζήσουν τη μητρότητα μόνες τους. Γιατί έχουν οικονομικές δυνατότητες και έχουν την επιθυμία έτσι να ζήσουν τη μητρότητα. Νομίζω λοιπόν ότι από πλευράς ε, Κοινοβουλίου θα πρέπει να προτείνουμε στοιχεία τα οποία να λαμβάνουν υπόψη την πραγματικότητα. Δεν μπορούμε να ορίσουμε κάτι πιο περιοριστικό από αυτό που υπάρχει στα κράτη-μέλη. Γι' αυτό νομίζω ότι θα πρέπει να εντάξουμε και άλλο τύπο οικογένειας που αναγνωρίζεται σε πολλές χώρες δεν μπορούμε να απομακρυνόμαστε από αυτή την πραγματικότητα ως προς τους ε, πατέ, προς τον πατέρα οι 19, 29 και 59 λαμβάνει υπόψη και τις ε, μονογονικές οικογένειες με μόνο τον πατέρα. Πολλές φορές ε, έχουμε να κάνουμε με ε, ζευγάρια από ομοφιλόφιλους και πολλές φορές δεν την χάνουν αναγνώρισης. Η κοινωνία δεν έχει τόσο υψηλή ανοχή. Γι' αυτό θα πρέπει να δούμε σε τι συμβιβασμούς πρέπει να φτάσουμε, γιατί πρέπει να συμπεριλάβουμε αυτές τις τροπολογίες και στο μέλλον να αναλάβουμε μία πρωτοβουλία όπου θα μιλάμε για άλλο τύπο οικογένειας, αλλά θα πρέπει να καταγράψουμε την κατάσταση και για τις μητέρες και για τους πατέρες. Προς αυτή την κατεύθυνση κινούνται οι τροπολογίες μας, διότι υπάρχει νομοθεσία, ειδική νομοθεσία σε ορισμένα κράτη-μέλη, την οποία δεν μπορούμε να αγνοήσουμε. Εμείς πρέπει να είμαστε οι εμπροστοφυλακοί που θα, αυτού που θα συμβεί στο μέλλον. Δεν μπορούμε να έχουμε μια περιοριστική οπτική γωνία. Και στο μέλλον μπορούμε να συντάξουμε μια έκθεση που θα λαμβάνει υπόψη και την άλλη αυτή πραγματικότητα. Ευχαριστούμε την κυρία Bilbao θα ήθελα να δώσω το λόγο στην κυρία Ματέρα, την εισηγήτριά μας. Ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ όλους και όλες που παρενέβησαν τις σκιώδης γιατί για εμάς αυτή θα είναι μία κοινή έκθεση. Θα πρέπει να είμαστε ενωμένες για την Ολομέλεια, διότι το θέμα είναι σημαντικό και τα στοιχεία είναι ε, δυστυχώς ανησυχητικά και ακολουθούν ανωδική πορεία. Συμφωνώ με Γκουρμάη ε, και Εστρέλα που μίλησαν για την μητρότητα και την πατρότητα. Πρόκειται για δύο όψεις του ίδιου νομίσματος και δεν πρέπει να γίνονται διακρίσεις. Όλοι έχουν τα ίδια δικαιώματα. Και αυτό αφορά και τον πατέρα που μεγαλώνει μόνος στο παιδί του, αν και είναι μικρή η ποσοστή αναλογία. Όμως θα πρέπει να ασχοληθούμε και με αυτούς, όχι όμως αυτή την έκθεση. Γιατί σας υπενθυμίζω αυτά που είπε η πρόεδρος Βένσεν. Ο, προ, ο τίτλος είναι σαφής. Ο τίτλος είναι απόλυτα σαφής. Χτες έγινε μία συζήτηση και με την κυρία Παρβανόβα. Και η κυρία Μπιλμπάου είπε ότι μπορούμε να εισαγάγουμε αυτή τη συλλογιστική στην αιτιολογική έκθεση ή σε να έχοντας υπόψη έτσι ώστε να μιλήσουμε και για αυτή την πραγματικότητα. Δηλαδή ε, ενός πατέρα που μεγαλώνει μόνο στο παιδί του. Αλλά τώρα μιλάμε για τις μητέρες, μιλάμε για γυναίκες. Εάν λοιπόν συμφωνείτε θα μπορούσαμε να ε, εισαγάγουμε αυτό το στοιχείο στην αιτιολογική έκθεση, αν και θεωρώ πολύ χρήσιμες τις τροπολογίες σας. Και η κυρία Παρβάνοβα μίλησε για την ανταλλαγή χρηστών πρακτικών, ανταλλαγή πληροφοριών για να καλύψουμε τα κενά. Θα λάβουμε υπόψη και αυτή την τροπολογία και συμφωνούμε και με μορφές πρόληψης, δηλαδή σεξουαλική εκπαίδευση στα σχολεία. Θα μπορούσαμε να λάβουμε υπόψη και αυτή την πτυχή. Κάτι που κάναμε. Αυτά είναι τα βασικά στοιχεία που θα πρέπει να μας απασχολήσουν για να υποβάλουμε μία έκθεση που να έχει νόημα, να είναι πλούσια, με συγκεκριμένα μέτρα που θα ληφθούν υπόψη και να λαμβάνει υπόψη όλες τις πτυχές. Γιατί αυτό είναι, αποτελεί την απαρχή της σκέψης μας. Θέλω να συμμεριζόμαστε όλοι τις ίδιες αρχές, όλες οι πολιτικές ομάδες και να ε, είμαστε ανοιχτές και σε συμβιβασμούς. Να βρούμε τις καλύτερες λύσεις που να είναι αποδεκτές από όλους. Έχω περισσότερο χρόνο από ότι για τον προϋπολογισμό, διότι θα ψηφίσουμε στις 15 Σεπτεμβρίου στο Στρασβούργο. Άρα όταν επαναλάβουμε τις εργασίες μας τον Αύγουστο θα έχω την δυνατότητα να ζητήσω μία συνάντηση των σκιωδών για να μιλήσουμε επί των θεμάτων και με όλες τις συναδέλφους που δεν είναι σκιώδεις αλλά θα θέλουν περαιτέρω διευκρινήσεις. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Ματέρα. Θα ήθελα να κάνω μία διευκρίνηση. Κατά τη διάρκεια αυτής της συζητήσεως ακούσαμε διάφορες απόψεις και ακούσαμε ότι η έκθεση αυτή μιλάει μόνο για τις ε, ε γυναίκες που μεγαλώνουν τα παιδιά τους μόνα τους. Ε, ε, μιλάει για τις μονογονικές οικογένειες και για τους πατεράδες που μεγαλώνουν μόνοι τους τα παιδιά τους. Αυτό ήθελα να διευκρινίσω και ε, χρειάζεται να έχουμε άδεια για να ε, καταρτήσουμε μία έκθεση. Ε, ε, γι' αυτό εμείς σε αυτή την έκθεση ζητήσαμε να αναφερθούμε μόνο για την κατάσταση των ε, ε, μοναχών μητέρων. Αν μιλούσαμε για μονογονικές ε, οικογένειες τότε θα είχαμε υπερβεί την εντολή που ανέλαβε αυτή η έκθεση και δεν θα μας επέτρεπα να καταρτήσουμε την έκθεση αυτή. Νομίζω ότι είναι σκόπιμο να σας υπενθυμίσω αυτό το γεγονός, γιατί τώρα έγινε μια ολόκληρη συζήτηση και ορισμένοι συνάδελφοι είπαν ότι η έκθεση αναφέρεται μόνο εις τις γυναίκες που μεγαλώνουν τα παιδιά τους μόνες τους. Υπάρχουν και άλλα θέματα τα οποία συζητήθηκαν σήμερα αλλά σας υπενθυμίζω ότι πρέπει να σεβόμαστε την εντολή που έχει δοθεί στην Επιτροπή μας. Η ψηφοφορία θα γίνει μέσα Σεπτεμβρίου και πριν κλείσουμε το θέμα αυτό της ημερησίας διάταξης, θα ήθελα να ευχαριστήσω και πάλι την ε, ε, εισηγήτρια για την ε, φιλοδοξία της, για τη συνεργασία της με τις πολιτικές ομάδες. Ίσως η κυρία Εστρέλα ήθελε να ρωτήσει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή εάν θέλει να σχολιάσει αυτό το θέμα. Δεν έχω έχουμε όμως χρόνο τώρα διότι η συζήτηση αυτή γίνεται μόνο για τις τροπολογίες. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα έπρεπε να παρουσιάσει τις θέσεις της κατά την πρώτη συζήτηση. Καλέψαμε λοιπόν τώρα αυτό το θέμα και έχουμε ακόμη μόνο ένα ακόμη σημείο στη μερίσια διάταξη την κατάσταση των θεμελιωδών δικαιωμάτων εντός Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Η συντάκτρια είναι η κυρία Σενκλέρ και ίσως καλό θα ήταν να πω στους συναδέλφους ότι δυστυχώς η κυρία Σανκλέρ σήμερα δεν μπόρεσε να έρθει εξού και αποφασίσαμε ότι θα ήταν ίσως καλύτερο να αναβάλουμε αυτή την έκθεση η οποία θα συζητηθεί στις 30 Αυγούστου όταν θα ξανασυναντηθούμε άρα μεταφέρεται και με αυτά φτάσαμε στο τελευταίο μας θέμα στα διάφορα. Δεν έχω ακούσει κανέναν να αναφέρει κάποιο θέμα στα διάφορα και η επόμενη συνεδρίμασή μας θα είναι στις 29 Αυγούστου και 30 Αυγούστου η κυρία Παπαδοπούλου όμως ζήτησε το λόγο. Κυρία Πρόεδρε, είμαι σκιώδης για την έκθεση αυτή της κυρίας Σανκλέρ και ήθελα να ξέρετε ότι για τις τροπολογίες έχουμε προσθεσμία ως τις 29 Αυγούστου. Αν τη συζητήσουμε λοιπόν την έκθεση 30 του μηνός, οι τροπολογίες θα έχουν τοποθετηθεί την προηγουμένη ε, και καλύτερα θα ήταν να το έχουμε συζητήσει. Είναι ένα ε, θέμα επουσιώδες, αλλά καλό θα ήταν να είναι εδώ η, η συγγήτρια διότι η ε, προθεσμία για τις ορπολογίες είναι για τις 29 του μηνός. Η κυρία Λούνατσεκ έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ την κυρία Παπαδοπούλου που έθεσε το θέμα αυτό, διότι και εγώ είμαι η συγγήτρια και ε, διαβάζοντάς το θα σας έλεγα ότι καλό θα ήταν να το συζητήσουμε τώρα διότι κατά τη γνώμη μου υπάρχουν πολλά θέματα που δεν αναφέρονται ή στη δικιά μας επιτροπή είναι θέματα ουσιαστικά για τα θεμελιώδη δικαιώματα εάν είναι ευρωπαϊκό δίκαιο ή διεθνές δίκαιο ή εθνικό δίκαιο χωρισμένα προβλήματα ε, λοιπόν, το να κατατεθούν τροπολογίες χωρίς να ξέρουμε τι θα αλλάξει η συγγήτρια είναι κάτι που θα μας δημιουργήσει πρόβλημα διότι μετά εάν θέλει να επιμείνει στις θέσεις που αναπτύσσει και ε, πιστεύω ότι δεν θα είναι μόνο η δική μου ομάδα η οποία θα έχει προβλήματα. Ίσως το πρόβλημα είναι της εισηγητρίας, αλλά ίσως ε, εάν ε, αναβάλουμε τη συζήτηση θα έπρεπε να αναβάλουμε και τις τροπολογίες. Ευχαριστώ. Κύριε Βεβαίως και πρόκειται να βρούμε μια ημερομηνία για τις ε, τροπολογίες. Αν δεν είναι η κυρία Σιγκλέρ, πώς θα ακούσουμε τις απόψεις οπότε. Θα πάμε για τις 30 Αυγούστου. Οπότε μπορούν όλες οι πολιτικές ομάδες και αυτόν τον τρόπο να υποβάλουν τις τροπολογίες τους. Στι, στις 2. 30 Αυγούστου, 2 η ώρα. Κύριε Παπαδοπούλου, έχετε λόγο. Κύριε Πρόεδρε, με όλο σεβασμό, νομίζω ότι αυτό δεν θα βοηθήσει και πάρα πολύ. Γιατί εάν γινόταν το πρωί η συζήτηση, θα πρέπει να εξηγηθεί από την συγγήτρια το πνεύμα της έκθεσης, η φιλοσοφία που διαπνέει το κείμενο. Οπότε ίσως να πρέπει να το κάνουμε το πρωί και να πάει η καταληκτική ημερομηνία αρχά Σεπτεμβρίου, ας πούμε 5 Σεπτεμβρίου η προθεσμία για τι τροπολογίε οπότε θα μπορέσουμε να ακούσουμε, παρακαλώ, <clears throat> θα ακούσουμε τις απόψει και θα ε, συζητήσουμε μετά. Ο Πρόεδρος. Ε, ε, συνάδελφοι θεωρούν ότι δεν θα καταφέρουμε να έχουμε τις ε, μεταφράσεις ε, για όλες τις ε, τροπολογίες, γιατί θα έχουμε μόνο στα αγγλικά τις τροπολογίες, επομένως θα πρέπει να παραταθεί η διάρκεια και η προθεσμία για τις τροπολογίες. Έχουμε και το θέμα βέβαια του ότι δεν είμαστε η αρμόδια της επιτροπή. Τέλο πάντων, να δούμε κατά πόσο μπορούμε να ε, μπορούμε να έχουμε ε, μια παράταση να πάει ας πούμε στις 5 ε, Σεπτεμβρίου το μεσημέρι. Επομένως, μεσημέρι της 5 Σεπτεμβρίου. Αγαπητοί συνάδελφοι, είμαστε στο 19 της ημερής διατάξεως. 29 και 30 Αυγούστου επομένω θα είναι η επόμενη συνεδρίαση και θα ήθελα να σα πω τα εξή πριν κλείσουμε τη συνεδρίασή μα. Πρώτα-πρώτα να ευχαριστήσω όλου του ε, συναδέλφου, όλου οι οποίοι ε, εργάστηκαν, οι οποίοι συνέβαλαν να ε, παράξουμε κάποιο έργο για τα δικαιώματα των ε, γυναικών και εγώ αισθάνομαι περήφανη με τιμά το ότι συνεργάστηκα μαζί σας ε, γιατί είσαστε αγωνίστριες ε, όλες έχετε συσπηρωθεί γύρω από αυτό το στόχο μας γύρω από το έργο μας και νομίζω για μένα ήταν μια υπέροχη εμπειρία το ότι συνεργάστηκα και επίσης βέβαια θα πρέπει να ευχηθώ σε όλους, σε όλες ε, καλές διακοπές, να ξεκουραστείτε, να, να, να, να ξεχάσετε ε, ε, και να φορτίσετε τις μπαταρίες και να έρθετε εδώ με πάρα πολλή ενέργεια. Επίσης πρέπει να ευχηθώ αντίστοιχα και στους συνεργάτες μας της γραμματείας. Μας διευκολύνουν πάρα πολύ το έργο. Επίσης, ευχαριστούμε και τους ε, διερμηνείς και εύχομαι σε όλους επομένως ευχάριστες καλές διακοπές. Θα τα πούμε επομένω μετά τις διακοπές τέλη Αυγούστου. Και θα συνεχίσουμε την διαδρομή μας όσον αφορά την ε, ισότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σας ε, ευχαριστώ και πάλι. Πέρα της συνεδριάσεως και όμως θα συνεχίσουν οι συντονιστές.